Συνάδελφοι, καθίστε αν θέλετε. Είναι ιδιαίτερα φορτωμένη η μερίσια διάταξη. Και κυρίω την έναρξη της συνεδρίαση. εφόσον συμφωνείτε. Je Παρακαλούμε να συγχωρήσετε τον κύριο Φερνάντε και του συναδέλφου από το ΕΛΚ, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συνέδριο στη Μαδρίτη, στο οποίο παρίσταται. Να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. και να σας ενημερώσω ότι η κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών ε, Προϋπολογισμών και ΛΥΜΠΕ θα οργανωθεί στις 27 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο στις 2 και 4 το μεσημέρι, 14 και 15. Θα ενημερωθούμε για, την, ε, για τον τριμερή διάλογο της 19ης Οκτωβρίου και μιας και ο Γενικός Εισηγητής λείπει, να πω εγώ ότι θύμισε τις τέσσερις πατριωτητές μας, τη δεσμεμέτρων για τους μετανάστες και πρόσφυγες, στα κεφάλαια 3 και 4, καθώς και τους οργανισμούς. Κατά δεύτερον, την αποκατάσταση των περικοπών στα προγράμματα 2020 και Connecting Europe Facility. εδώ και αυτό θύμιζε ο κ. Φερνάντες ότι δεν θέλουμε να διακοπούν οι πρωτοβουλίες για την απασχόληση των νέων και τέλος τέταρτη προτεραιότητα ή στόχος ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσεις στα πλαίσια του πολιτού προγραμματισμού των πληρωμών και κυρίως να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία ευελιξία που προβλέπονται στο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου ο Υπουργό του Λουξεμβούργου μας θύμισε ότι υπάρχει μια πέμπτη προτεραιότητα που ήταν να γίνουν σεβαστές οι οροφές, τα ανώτατα όρια του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Υπογράμμισε ότι έχουμε κάποιες εγγραφές αρνητικές και αυτό προϊονίζει την ε, συνδιαλλαγή που θα είναι μάλλον απατητική και ίσως και ιδιαίτερα δυσχερής. Κατόπιν αυτών, να δώσω το λόγο στον εισηγητή μας για τα υπόλοιπα τμήματα, τον κύριο Ντεπρέ, και μετά στον κύριο Γκάγερ για τους οργανισμούς. Και ο ένας και ο άλλος συμμετείχαν στον τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σχετικά σύντομος. Θύμησα τις επιλογές που είχαν γίνει από την Επιτροπή Προπολογισμών για τα υπόλοιπα τμήματα και επειδή τα έχουμε ήδη ψηφίσει δεν χρειάζεται να επανέλθω. Το μόνο σχόλιο που έγινε από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου αφορούσε την μείωση του προσωπικού 5% μείωση αναπόσπαστο τμήμα του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου επέμεινε ιδιαιτέρως στο να γίνει σεβαστό από όλα τα θεσμικά όργανα το όριο αυτό. Σε αυτό απήντησα ότι υπάρχει ε, διαφορά στην ε, αποτίμηση του όλου θέματος από εμάς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κυρίως ε, την περίμετρο, το πλαίσιο το οποίο θα εφαρμοστεί αυτό το ποσοστό. Ε, πρέπει λοιπόν στο επίπεδο της συνδιαλλαγής να προσέξουμε αυτές τις ευαίσθητες διαπραγματεύσεις για να περάσει και η δική μας άποψη για τις θέσεις του Συμβουλίου. και να υπερασπιστούμε τη θέση μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Άρα επιμείνατε στο ότι το Κοινοβούλιο σέβεται τις υποχρεώσεις του. Πρόεδρε, σε αυτή την φάση δεν προσπάθησα καν να πείσω. Απλώ εξήγησα ότι υπάρχει διαφορά στην αποτίμηση. Δηλαδή θα πρέπει να διαπραγματευτούμε με ιδιαίτερη πυγμή για το θέμα αυτό. Δεν είναι προσωπική μου άποψη. Σα εξήγησα βάση των ψηφοφοριών στην Επιτροπή Προπολογισμών τι εντολή έχω εκ μέρου του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε κύριε Γκάγερ για του οργανισμού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο κι εγώ. Το σκεφτικό μου ήταν στο πλαίσιο του πρώτου τριμερούς διαλόγου το είχα πει στην ε, Προεδρία του Συμβουλίου. Προσπαθήσαμε δηλαδή να κάνουμε κάποιες τεχνικές συνεδριάσεις για να ασχοληθούμε με όλα εκείνα τα ζητήματα τα οποία μπορούσαν να χωριστούν από την κύρια διαπραγμάτευση. Είναι ακόμα ανοιχτό το θέμα το αν θα δεχτεί κάτι τέτοιο η Προεδρία, θα το αποφασίσουν η Λουξεμβουργική Προεδρία, φαντάζομαι όχι μόνη της, δεν ξέρω αν θέλουν να δεχτούν αυτή την προσφορά, εάν όχι... Οι διαπραγματεύσει για αυτό το πολύ μικρό τμήμα του προπολογισμού θα πέσουν μαζί με το υπόλοιπο. Βεβαίω το μεταναστευτικό πακέτο δεν μπορούμε να το δούμε χωριστά από τον προπολογισμό και το προσωπικό της Frontex, της EASO και της Europol βεβαίως. Αλλά μπορεί να μας διευκολύνει αυτό το οποίο είπα και πρότεινα και θα δούμε τώρα το αν θα δεχτεί την προσφορά μας στο Συμβούλιο. Μια παρατήρηση για τις διαπραγματεύσεις. Ήταν σωστό και εμείς επιμένουμε στη θέση μας όσον αφορά τον ρόλο των ε, μέσων στο πλαίσιο του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου που, έχουμε στην, ε, που ψηφίσαμε στην πρόταση περιπολογισμού. Αλλά το εάν μπορεί να αφήσει πίσω του αυτά τα οποία είχε ως ιδέες για το πολιτισμό δημοσιονομικό πλαίσιο το Συμβούλιο δεδομένων των μεγάλων προκλήσεων ε, δεν ξέρω, αμφιβάλλω. Δεδομένης ε, κυρίως της πίεσης από τα κράτη-μέλη. Και εκεί ήταν σαφής η Προεδρία. Θυμάμαι μάλιστα χαρακτηριστικά είπαν πως ε, άλλο πράγμα η χρηματοδότηση και άλλο η δημοσιονομική πειθαρχία. Οπότε βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση να προχωρήσουν πέρα από το υπάρχον δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε λοιπόν αυτές τις τροποποιητικές επιστολές της ε, Κομισχέων ε, που μειώνουν ακόμη περισσότερο το περιθώριο που υπάρχει ακόμα και για δεκαδικά ψηφία μιλάμε. Ε, κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό. Όχι εδώ, κάπου θα πρέπει να γίνει όμως, κάπου θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ο τριμερής αυτός διάλογος ε, ήταν, αν θέλετε, κάποιο είδους ε, συνάντηση για να υπάρξει μια συνδιαλλαγή και βεβαίως έχουμε και την, ε, το, το σχέδιο προπολογισμού του 2016. Λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι πως σαφώς ο προπολογισμό αυτός δεν θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει για το 2016 αλλά και τις προκλήσεις ε, το μεταναστευτικό κάτι το ναι. οποίο δε, από ό,τι φαίνεται δεν θα μειωθεί ξαφνικά κάθε άλλο πρέπει λοιπόν να βρούμε τους πόρους που χρειαζόμαστε για ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και ίσως να υπάρξει και εκεί πέρα μια μεγάλη ε, παρέμβαση για να επιτρέψουμε και κάποια, και κάποια ανάπτυξη στην υποσαχάρη Αφρική και για να υπάρξει κάποια επιστροφή των ανθρώπων που είναι τώρα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις πατρίδες τους. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια εντύπωση, αλλά νομίζω πως ο προπολογισμό μας ναι. ε, σε σχέση με τις δεσμεύσει που έχουν αναλάβει οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και ως προς τις δηλώσεις που έγιναν, νομίζω ότι ο προπολογισμό αυτό δεν είναι στο ύψο των ε, υποχρώσεων που μας περιμένουν να φέρουμε ει πέρα. Νομίζω λοιπόν ότι στη συνδιαλλαγή θα έχουμε πραγματικά σοβαρές δυσκολίε και θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να φανούμε ιδιαίτερα διαλλακτικοί, να δείξουμε κατανόηση και θα είναι πραγματικά φοβερή η δοκιμασία. Ας παραμείνουμε σε αυτά ως προς την ε, έκβαση του πρώτου τριμερού διαλόγου. Τώρα, για τη δεύτερη διευθυντική επιστολή μας έχει ήδη να αλλά να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής για τα βασικά χαρακτηριστικά της. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία της διορθωτικής επιστολής. Την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε αυτό το, το, πάγιο γράμμα, αυτή την ε, επιστολή σε σχέση με τις ε, δαπάνες. Υπήρξε επομένω κάποιο είδους ενημέρωση και έτσι τώρα θα έχουμε προγνωστικά πιο ασφαλή και ακριβή για χρόνο Υπάρχει όμω και ένα άλλο τώρα ε, καινούριο στοιχείο σε αυτή τη διορθωτική επιστολή. Πρόκειται για τις επιπτώσεις του προϋπολογισμού σε σχέση με τα πιο πρόσφατα πακέτα που έχουν ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο. Και έτσι θα αντιμετωπιστεί το μεταναστευτικό και η κρίση λόγω της ροής των προσφύγων. Οπότε για να ξεκινήσουμε αυτή τη γενική έποψη και μετά να δούμε τα επιμέρους θέματα. Πρώτα-πρώτα για να δούμε τι γίνεται με τη δέσμη μέτρων για το μεταναστευτικό. Γενικώ σε αυτή την τροποποιητική επιστολή προτείνει η Επιτροπή να ενισχυθούν τα μέτρα τα οποία αφορούν το 1,5 δις από τις επιστώσεις υποχρεώσεων. Και αυτό θα έχει να κάνει με την κρίση των προσφύγων και θα γίνει αυτή η αύξηση κατά ένα ακόμα δις για τις πιστώσεις υποχρεώσεων. Αυτό περιλαμβάνει και 140 εκατομμύρια, τόσο ώστε να αυξηθούν οι πιστώσεις για την ανθρωπιστική βοήθεια, ούτως ώστε να καλύψουμε τις πιο επίγουσες ανάγκες της τρίτης χώρας και ιδίω στις γειτονιάζουσες. Στο κεφάλαιο υπαριθμών 3 υπάρχει μια δεσμή μέτρων. Θα σας πω σε λίγο και εκεί αυξάνονται οι δαπάνες της πιστώσης υποχρεώσεων κατά 1 δις 380 εκατομμύρια και 779 στις πιστώσει πληρωμών 379 εκατομμύρια οπότε έτσι έχουμε την πρώτη δεσμή μέτρων όσον αφορά την ενίσχυση της κατεπηγούσης αροχής για το Ταμείο για Άσυλο και Μετανάστευση. Και επίσης όσον αφορά το Ταμείο για την Ασφάλεια και αυτή η δεσμή μέτρων αντιστοιχεί σε 94 εκατομμύρια σε πιστώσει υποχρεώσεων. Έχουμε τώρα μια δεύτερη δεσμή μέτρων που αποσκοπεί στο να καλύψει τις δαπάνες όσον αφορά την επανεγκατάσταση και τα σχετικά μέτρα. Έχουμε δύο διαφορετικές ε, αποφάσεις του Συμβουλίου για την επανεγκατάσταση. Ξεκίνησαν με 40.000 πρόσωπα οι οποίοι θα επαναγκαθίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ακολούθησε δεύτερη δέσμη για άλλους 120.000. Άρα συνολικά έχουμε 160.000 πρόσωπα τα οποία θα επανακατασταθούν και οι σχετικές ε, πιστώσεις που προτείνονται για το 2016 συνολικά ανέρχονται στα 890 εκατομμύρια πιστώσεων για το 2016. Μία τρίτη μέτρων αφορά την Frontex. Εκεί έχουμε μία αύξηση 70 εκατομμυρίων όσον αφορά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της Frontex. Ιδίως δε όσον αφορά την επιστροφή σε σχέση με τη συνεργασία με τα κρατη όσον αφορά επίσης την ε, ε, έναρξη λειτουργίας των κέντρων καταγραφής, των hotspots. Και εδώ έχουμε τον δεκατομμύριο Τώρα, μια τέταρτη δεσμή είναι η αναβάθμιση των τριών υπηρεσιών της πρώτης γραμμής, Frontex, EASO και Europol. Και εκεί έχουμε την αύξηση προσωπικού τους και για τις τρεις υπηρεσίες είπαμε να γίνει αύξηση συνολικά 120 θέσεων. Και το 2016 είπαμε ότι θα είναι πλήρως λειτουργικέ αυτές οι υπηρεσίες και το δε υπολογίζεται σε περίπου 16 εκατομμύρια για τις τρεις αυτές υπηρεσίες. Τέλος, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία αύξηση 310 εκατομμυρίων για το για το άσυλο δηλαδή αλλά και για το ΆΜΕΦ που έχει σχέση με τον επαναπατρισμό, 48 εκατομμύρια και επίσης για το Ταμείο Ασφάλειας των Ιστορικών Συνόρων που έχουμε και αύξηση 82 εκατομμύρια. Έτσι θα αναβαθμιστεί η υποδοχή των, ετούντων άσυλων. Γιατί η είναι χωρίς προηγούμενο και επίσης έτσι θα γίνει και η διεκπαιρέωση των αιτήσεων ασύλου. Με αυτόν τον τρόπο εν μέρη θα καλύψουμε τις ανάγκες από την μεταναστευτική πίεση και τα όσα χρειάζεται να γίνουν στα εξωτερικά σύνορα. στο κεφάλαιο 3 είπαμε ότι φτάσαμε στην οροφή για το 2016. Οπότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να ενεργοποιήσουμε το εργαλείο ευελιξίας κάτι το οποίο προβλέπεται από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε και συνολικά θα καλύψουμε τα 124 εκατομμύρια τα οποία ήδη προέβλεπε το σχέδιο προπολογισμού για το όργανο ευελιξίας. Οπότε συνολικά πάμε στα 1,5 δις τα οποία θα εκταμιευθούν με το, όργανο, με το εργαλείο ευελιξίας ε, σε σχέση με την οροφή του κεφαλαίου παρθμών 3. Να σας δώσω τώρα τη, μια ιδέα της τάξης μεγέθους αυτής της προσπάθειας που γίνεται για την εκταμίευση όλων αυτών των κονδυλίων για το 2015 και 2016 το ποσό των κονδυλίων που θα εκτομιευθούν φτάνουν στα 9,2 δις. Δηλαδή δύο φορές περισσότερα από όσο αρχικά είχαν προγραμματιστεί για τα μέτρα του κεφαλαίου 3 και 4 για να καλυφθεί η πρόληψη, πρόληψη του μεταναστευτικού. Επίσης αυτά τα 9,2 πρόκειται να καλύψουν και το καταπίστευμα για την Αφρική. Εκεί όπου κάποιοι από αυτού του πόρου θα προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Για να δούμε τώρα τι γίνεται όσον αφορά την γεωργία. Τι προβλέπει δηλαδή η διορθωτική επιστολή που είναι ε, κάτι το οποίο παραδοσιακά φύγεται ε, σε αυτή τη διορθωτική αποστολή εδώ. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναβαθμίσουμε και να ενισχύσουμε τα 50 μέτρα. Μιλάμε για 700 εκατομμύρια. Από τα, 500, από τα 700 τα 500 θα είναι κάποια προσωρινά μέτρα στα γαλακτοκομικά και ε, λίγα χρήματα για το χείριο κρέας. Επίσης θα έχουμε για προκυβευτικά κάποια μέτρα στήριξης όπως αποφασίσουμε από μερικούς μήνες κατόπιν της παράτασης ε, του εμπάργου της Ρωσίας για τις ε, εισαγωγές. Οπότε σε σχέση με το σχέδιο προπολισμού του 16 του τέλους Μαΐου έχουμε αύξηση για αυτές τις δαπάνες. Αύξηση κατά 700 εκατομμύρια. Τώρα όσον αφορά τις ε, στόσεις υποχρεώσεων για το 2016 και εδώ είναι καλά τα μαντάτα ότι δηλαδή το, τα, τα έσοδα τα οποία θα προέλθουν από τις επιβαρύνσεις στο γάλα και την εκαθάριση των λογαριασμών θα είναι επίσης ε, λιγότερο από όσο περιμέναμε η απορρόφηση το 2015. Άρα αυτά τα έσοδα τα οποία θα καλύψουν μέρος των εξόδων θα φτάνουν το 1,1 δις παραπάνω από όσο αρχικά είχε προβλεφθεί όταν συντάσαμε το σχέδιο προπολογισμού και καθαρή επίπτωση των αυξήσεων των δαπανών όπως προτείνονται για αυτά τα διαθέσιμα έσοδα σημαίνει ότι μπορούμε να προτείνουμε κάποιες πιστώσεις για το Ταμείο Γεωργικών Εγγύσεων. Μιλάμε 477 εκατομμύρια κάτω από όσα προέβλεπε το σχέδιο προπολογισμού για το 2016. Παρά αυτά, το σύνολο της δαπάνης για την ε, γεωργία παρουσιάζει αύξηση 660 εκατομμύρια σε σχέση με την αρχική πρόταση. Την ε, τροποποιητική διορθωτική επιστολή επίσης έχουμε και άλλες προτάσεις. Να σας τις πω εντάχει. Πρώτα πρώτα έχουμε αύξηση 5 εκατομμυρίων. Έτσι θα καλύψουμε κάποιες υποχρεώσεις σε σχέση με το Ταμείο Επενδύσεων και έτσι θα γίνει και η εκτέλεση του προγράμματος του Ταμείου για τις ΜΜΕ και θα αφορά προγράμματα ε, σύμφωνα με το Ταμείο για Στατικές Επενδύσεις αυτό θα έχει προσωρινό χαρακτήρα γιατί και στη συνέχεια αυτό το παράθυρο πρόκειται να καλυφθεί από τους χρήστες για τα επόμενα χρόνια. Επίσης, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιες μειώσεις στον αφορά τον υπολογισμό των δαπανών για τις αλληλευτικές διεθνείς συμφωνίες αλλά και για το πρόγραμμα που αφορά τα είδη διατροφής και επίσης τα ε, κτηνοτροφές σύμφωνα με τις προβλέψεις των δαπανών. Επίσης προτείνει η Επιτροπή αύξηση 23 εκατομμύρια των πιστώσεων για αμοιβή του, αμοιβές του προσωπικού. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έχει τις θέσεις υπαλλήλων όπως προβλέπονται από το πρόγραμμα που προέβλεπε 1% αύξηση θέσεων. Και κατά αυτόν τον τρόπο τώρα είπαμε ότι θα έχουμε μέσο όρο κενών θέσεων 3,4%. Αλλά θα εξυπηρετηθεί και ο στόχος του 5% για μείωση. Όμως έτσι κάποιες κενές θέσεις μπορούμε να τις ε, αναθέσουμε σε κάποιους πιο αποτελεσματικά. Και έτσι τελικά για όλη τη χρονιά κατά μεσοσταθμικά θα έχουμε λιγότερες χειρεύουσες θέσεις. Αυτά όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών που θα χρειαστούν κυρίως για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό αλλά επίσης ε, και ότι υπάρχει ανάγκη να αναβαθμίσουμε κάποιες υπηρεσίες της Επιτροπής που δρούν στην πρώτη γραμμή σε αυτό το μέτωπο. Τέλος, η διορθωτική επιστολή προτείνει και κάποιες τεχνικές προσαρμογές όσον αφορά το πρόγραμμα για την ε, υπηρεσία συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας. Και κάποιες λοιπόν προς μικρές προσαρμογές και αλλαγές του προγράμματος. Αυτά και είπαμε ότι συνολικά όσον αφορά τις δαπάνες, σύμφωνα με την επιστολή έχουμε αύξηση ένος της 70 εκατομμυρίων όσον αφορά τις πιστώσεις υποχρεώσεων για το 2016. Και όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών έχουμε αύξηση 914 εκατομμύριων. Ελπίζουμε ότι αυτά τα στοιχεία της διορθωτικής επιστολής θα ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της συναλλαγής και επίσης θα συνεχίσουμε ε, αυτή την θετική ε, παράδοση των 7 ε, διορθωτικών προπολογισμών στα τους οποίους τα έχουμε βρει μέχρι τώρα. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε κύριε Φεζά για αυτήν την ε, παρουσίαση. Καταλάβαμε λοιπόν ποια είναι η ουσία, οι αδρές γραμμές της διευθυντικής επιστολής παριθμών 2. Σε ένα βαθμό τα είχατε προβλέψει από την Επιτροπή. Βεβαίω όλα αυτά θα καλυφθούν πλήρως μόνο κατά τέτοια συμβιαλλαγή. Ε, ο κύριος Ντεπρέ έχει ζητήσει το λόγο ή ο κύριος Γκάγερ. Είχα σημειώσει τον κύριο Ντεπρέ. Όχι, πρόεδρε, νομίζω ο εισηγητής για την ομάδα του για την ερχόμενη χρονιά είναι ο κύριος Γκάγερ. Οπότε του παραχωρώ το λόγο. Για λόγους προτεραιότητας. Ναι, δεν είχα ζητήσει το λόγο. Αλλά βέβαια αφού μου το δίνετε, τι να κάνω κι εγώ. Κοιτάξτε, αφενός έχουμε τροπολογίες οι οποίες ε, απλά προσπαθούν να εφαρμόσουν στο πεδίο του προπολογισμού τις πολιτικές αποφάσεις όσον αφορά δηλαδή τις αποφάσεις μετεγκατάστασης Αυτό είναι το οποίο το στηρίζουμε βεβαίως ως κοινοβούλιο είναι μια σημαντική πολιτική απόφαση αλλά και χρειάζεται βεβαίω και κονδύλια για να εφαρμοστεί. Και δείχνει βεβαίω, ακόμη μια φορά πως ε, αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι περισσότερα από όσα προέβλεπε μέχρι τώρα το σχέδιο προπολογισμού της Κομισιόν και του Συμβουλίου. που είχαν μείνει στα δεδομένα του καλοκαιριού. Οπότε θα πρέπει σε τελική ανάλυση το Συμβούλιο να αναγνωρίσει ότι δεν γίνεται, άμα παίρνει στα σοβαρά αυτά τα οποία λέει, να συνεχίσει να εργάζεται με αυτή την πρόταση προπολογισμού. Βεβαίω ε, αναμένουμε κι εμεί κάποια ένδειξη πότε θα έρθει το Συμβούλιο με μια πρόταση που θα είναι προσαρμοσμένη στα γεγονότα. Γιατί μόνο τότε μπορεί να ξεκινήσει σοβαρή διαπραγμάτευση. Γιατί ε, βλέπετε ότι δεν συμβάζεται με την πραγματικότητα. Έχω τώρα μια μικρή ερώτηση για ένα δευτερεύον ζήτημα. Ε, μου προξενεί κάπως έκπληξη για το ότι η Κομισιόν ε, θεωρεί υπεύθυνη τη Frontex ε, για τις επιστροφές. Μέχρι τώρα αυτό είναι αρμόδια των κρατών μελών, αρμοδιότητα των κρατών μελών. Σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, αν κάποιος ε, δεν ε, έχει καθεστώ ε, πρόσφυγα, τον οδηγεί η αστυνομία στο αεροδρόμιο και το πληρώνει το γερμανικό κράτο. Τώρα χωρίς να είμαι ειδικό στο θέμα και να γνωρίζω ακριβώς την θεωρία, αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί θεωρητικά κάποιο κράτος μέλος να πει εντάξει θα πάρω τα λεφτά αυτά για να πληρώσω τους επαναπατρισμούς. Θεωρητικά, εντάξει, ναι. γίνεται. Δεν ξέρω πόσο έξυπνο είναι. Ξαφνικά μια εθνική αρμοδιότητα να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ στο πλαίσιο της επικουρικότητας το θεωρώ λάθος, αλλά τέλος πάντων η κατάσταση τώρα έχει έτσι που δεν έχει νόημα να επιμείνουμε σε αυτό το ζήτημα αρχής. Αλλά γιατί τη Frontex. Εντάξει, ε, το νόημα του να έχουμε μια υπηρεσία είναι να αναλάβει πραγματικά κάποιε αρμοδιότητε που ήταν των κρατών μελών. Αλλά οι επαναπατρισμοί δεν είναι αρμοδιότητα. Οι επιστροφέ δεν είναι αρμοδιότητα τη Frontex. εκτός να τις δώσουμε αρμοδιότητα και μετά ξανασυζητήσουμε τον προϋπολογισμό και το προσωπικό της. Γιατί τι γίνεται. Ε, αναθέτει η Κομισιόν, αναθέτει η Ένωση σε κάποιες ε, τέτοιες υπηρεσίες, κάποιες αρμοδιότητες και μετά λέει για αυτές τις αρμοδιότητες χρειάζονται αυτά τα μέσα. Δηλαδή αυτό δεν έχει γίνει τώρα μια τέτοια αιτιολόγηση μέχρι στιγμής. Είναι, είναι δύσκολη η κατάσταση. Για αυτό το συγκεκριμένο σημείο, εγώ κατάλαβα ότι για, το hot για τα hot spot ήταν το θέμα των επιστροφών. Έτσι είναι κύριε Ντεπρέ. Πρόεδρε, αν θέλετε να απαντήσω στην ερώτηση τώρα ή μετά. Ε, μετά, ε, μετά. Μπορείτε να απαντήσετε μετά το άλλο θέμα. Η κατάσταση είναι περίπλοκη, ειδικά αυτή τη στιγμή, γιατί Δευτέρα βράδυ μας είπε το Συμβούλιο, είναι σημαντική η δημοσιονομική πειθαρχία, κατέθεσε τον 8ο τροποποιητικό προπολογισμό η Κομισιόν, έριξα μια γρήγορη ματιά εγώ στα νούμερα και αυτό τα νούμερα σημαίνουν ότι ευτυχώς ε, υπάρχουν 9,8 δισεκατομμύρια επιπλέον έσοδα από τα, ε, τους ίδιους πόρους. Όχι 9,4, λάθος. τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν το αντιλαμβάνομαι σωστά οι εκτιμήσεις ε, της Κομισιόν ε, ήταν μέχρι στιγμής πάρα πολύ απεσιόδοξες ή συντηρητικές εάν θέλετε καθώς εισέπραξε 9,4 δισεκατομμύρια παραπάνω από όσο προϋπολόγιζε τώρα αυτά είναι ε, στην διάθεση των ε, κρατών μελών, κάτι για το οποίο βεβαίω χαίρονται οι Υπουργοί Οικονομικών και των 28 κρατών μελών. τι θα κάνουμε τώρα με αυτά τα λεφτά θεωρητικά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτήσουμε περαιτέρω δραστηριότητες, ε, οπότε το επιχείρημα που μας είπε το Συμβούλιο Δευτέρα βράδυ περί δημοσιονομικής ε, είναι λίγο πιο ασθενές πλέον. Ε, υπάρχουν διάφορα δόγματα, αντιλαμβάνομαι βεβαίω γιατί χρειάζεται ακριβώς το πλαφόν στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και αντιλαμβάνομαι πως υπάρχει Μεγάλη Βρετανία και είναι ιδιαίτερο σκληρό το δόγμα αλλά δεδομένου του ότι είχαμε ανέλπιστα υψηλά έσοδα νομίζω πως ε, ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη στην πολιτική μας σκέψη. αυτό και θα ήθελα να ακούσω κάποιες ε, δικές σας σκέψεις για αυτά τα 9,4 δισεκατομμύρια. Ευχαριστώ. Κύριε Ντεπρέ, ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτη μου παρατήρηση, χαίρομαι από το Κοινοβούλιο σε αντίθεση με το τι γίνεται συνήθως για την πρόταση αύξησης πιστώσεων και στις αναλήψεις υποχρεώσεων και στις πληρωμές, όπως πρότεινε η Επιτροπή Προπολογισμών και όπως τώρα προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Διευθυντική Επιστολή Περιθμών 2, ε, πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση, ακόμη και αν υπάρχουν κάποιες μικρές αποκλήσεις στην ε, εκτίμηση των απακριβών ποσών. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι τουλάχιστον συμφωνούμε και είμαστε ενωμένοι ως προς την άλλη αρχή του προπολογισμού Δημοσιονομική Αρχή για το τι πιστώσει χρειάζονται. Αυτό ισχύει για το κεφάλαιο 3 και για το κεφάλαιο 4, κυρίω για την αύξηση τη ανθρωπιστική βοήθεια και ισχύει και για την ενίσχυση των πιστώσεων στα θέματα γεωργία. Να εκφράζω λοιπόν την ικανοποίησή μου και ελπίζω ότι η ένωση των δυνάμεών μα θα δώσει θετικά αποτελέσματα. Έχω όμως κάποια ερωτήματα προς τον κύριο και τον, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις, στο τμήμα 3, στις πιστώσεις που προτείνεται, για την ε, επανεγκατάσταση 120.000 άτομα προτείνεται να καλυφθούν από τα, τα ταξιδιωτικά τους. Τα 500 ευρώ όμως ε, για τα οδηπορικά αφορούν τις 120.000, όχι τα πρώτα 40.000 που πρόκειται να επανακατασταθούν. Αυτό καταλαβαίνω από το σημείωμα. Εάν λοιπόν για τους 120.000 προβλέπονται 500 ε, οδηπορικά να <clears throat> γιατί οι 40.000 πρώτοι δεν επωφελούνται από αυτό το ποσό, γιατί αυτή η διαφορά. Δεύτερη ερώτηση. Και ξανάρχομαι σε ένα θέμα που ήδη μας έχει απασχολήσει προηγουμένω. και έχει να κάνει και με τις παρατηρήσεις του κυρίου Γκάγερ για την Frontex. Είναι σαφές το ανακοίνωσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι σκοπεύει στην Frontex να δώσει δικαίωμα πρωτοβουλίας για την διοργάνωση του κόστους. Το δικαίωμα της πρωτοβουλίας αυτή τη στιγμή δεν το έχει. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει συζήτηση για την ε, τροποποίηση της νομικής βάσης που το επιτρέπει. Όμως, με ευνηδιάζει και σε αυτό είχαμε επιμείνει στο παρελθόν, το τι θα γίνει με τη βάση που έχει να κάνει με τις επιστροφές. Τα 38 πρόσθετα εκατομμύρια που ζητάτε για τις αναλήψεις πληρωμών και τα 17 για τις πληρωμούς κυρίως θα τα πάρουμε από την ε, ε, δημοσιονομική γραμμή 18.03.01.02 και ο τίτλος της είναι αρκετά ε, ιδιαίτερος. Η προώθηση των, ε, των ε, δραστηριοτήτων για τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ένταξη των υπηκών τρίτων χωρών με μια συγκεκριμένη στρατηγική. Δηλαδή η ίδια δημοσιονομική γραμμή χρησιμοποιείται ταυτόχρονα για να πούμε ότι θα προωθήσουμε την ένταξη των υπηκών τρίτων χωρών και ταυτόχρονα για την ε, επανακατάστασή τους. Είναι κάπως περίεργο. Γιατί στην προηγούμενη συζήτησή μας λέγατε ότι δεν είναι εύστοχο να αλλάξει ο τίτλος του ταμείου. Το ταμείο για τους πρόσφυγες. τρίτη ερώτηση η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χρηματοδότηση του Ταμείου Μαντάτ. το οποίο θα ενισχυθεί με πιστώσεις της Ένωσης και με εθνικές συνεισφορές. Στον προπολογισμό όσο έχει αυτή τη στιγμή με τη διορθωτική 2 έχετε τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα για να το καλύψετε και ως προς τα ποσά που είχαν αρχικά αναγγελθεί. Νομίζω, επειδή δεν είμαι βεβαίως, ότι θα μπορούσατε να μας το επιβεβαιώσετε. Και τελευταία ερώτηση. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που αυτή τη στιγμή βρισκόνται σε εξέλιξη με την Τουρκία. Αρχικά μιλούσαμε για ένα δις ευρώ επιπλέον ποσό. Η Τουρκία ανεβάζει λίγο το ποσό ε, και αν δεν υπάρξουν τρία δι, δεν φαίνεται να, προ... να διαφαίνεται συμφωνία. Και αν κατάλαβα καλά τι τουρκικέ θέσει, τρία δι για όσα γίνονται στο επίπεδο των ε, πιστώσεων προενταξιακά. Αυτά τα τρία δι ευρώ. Και εφόσον υπάρξει συμφωνία με την Τουρκία, από πού θα βγουν. Πού θα τα βρούμε, από πού θα τα εκταμιεύσουμε. Θα επιβαρύνουν τον προπολογισμό το 2016. Θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερη μέθοδος ε, χρηματοδότηση. Δηλαδή, πιο ξεκάθαρα, θα πρέπει να περιμένουμε αύξηση των πιστώσεων κατά 3 δις για το 2016, για τον προβλεπόμενο του 2016 και για την ε, προβλεπόμενη συμφωνία με την Τουρκία. Ευχαριστούμε κύριο late So the... Ευχαριστώ. Ε, έχασε ένα μέρος του τόσο θετικού μηνύματος χαράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, αλλά κάποια θέματα νομίζω πρέπει να τα δούμε καλύτερα. Έχω την αίσθηση είναι πολύ περίεργο το παιχνίδι της Επιτροπής ε, για να καταλήξουμε στο διαμηδενικό αποτέλεσμα. Μόλι προτείνουν κάτι θετικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη θα επανέλθουν με κάτι λίγο πιο αρνητικό και τελικά θα καταλήξουμε στο μηδενικό αποτέλεσμα. Όπως άλλοτε ακούγοντα του αριθμού που αναφέρθηκαν, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τα διαφορετικά προβλήματα του μέλλοντο που τα έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρξει πραγματική διόρθωση. Θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την... Ε, το αποθεματικό. Αυτή είναι η βασική μου ερώτηση. Κατά τα άλλα, καταλαβαίνω ότι ο γαλακτοπαραγωγικό τομέα και το χείριο θα πάρουν τα ποσά που του αναλογούν. Και αυτό είναι ένας κίνδυνος που θα μπορούσε να ε, αντιμετωπιστεί αν ε, προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει το ρωσικό Εμπάργκο. Κάπου πριν από δύο μέρες διάβασα ότι πληρώνουμε πάρα πολλά για την αλία. Και είδα ένα φρικτό ποσό, κάτι σαν 600 εκατομμύρια. Σε κάποια φάση ήμουν σκιώδης για κάποιες εξελιχτικές συμφωνίες. Και νομίζω ότι είχα δίκιο τότε όταν έλεγα ότι αυτά συμβαίνουν Μάλλον τυχαίνει καμιά φορά να έχω και δίκιο και έλεγα τότε ότι είναι πολύ δαπανηρές οι συμφωνίες αυτές. Τώρα έχουμε ένα, μια λυπητερή στα χέρια μας, τρομερή, και καλό θα ήταν να έχουμε κάποιες διευκρινήσεις προς αυτό. Ευχαριστούμε κύριος Μαραγκάλ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος, θέλω να ρωτήσω ακριβώ το ίδιο, όπως και ο κύριο Ντεπρέ. Τι γίνεται με την συμφωνία με την Τουρκία. Και να σας πω και μία σκέψη μου. Αυτή τη βδομάδα είδαμε η κυρία Μέρκελ να φέρεται και σαν πρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σαν πρόεδρο του Συμβουλίου και σαν καγκελάριο της Γερμανίας. Υπέροχο καθισμένη στο παλάτι του κυρίου Ερντογάν, στο θρόνο. Οπότε υπ' αυτές τις τρεις ιδιότητες μπας και μπορεί να λύσει και το δημοσιονομικό πρόβλημα. Πάντως εμένα με ανησυχεί κάτι. Νομίζω ότι είναι λάθος το να αντισταθμίζεται η ισορροπία που θα πρέπει να υπάρχει ε, σε αυτή τη συμφωνία για τους ε, πρόσφυγες και να αντισταθμίζεται αυτό και να εξισορροπείται με το κόστος της προένταξης. Νομίζω ότι αυτό από πλευρά τη είναι πάρα πολύ συζητήσιμο. Επίσης, κάτι άλλο για τη γεωργία. Να σας πω ότι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα βλέπουμε ότι βρισκόμαστε σε θέση κάποιου διαχειριστή που κάνει, έχει ρόλο αναδιανεμητικό. Όμως θέλαμε μια αναδιάρθρωση της γεωργίας. Και αυτή η ανάγκη για μεταρρύθμιση γίνεται όλο ένα και πιο επιτακτική. Ευχαριστώ κύριο. Πρόεδρε. Άκουσαν ήδη πολλά επιχειρήματα. Είναι κρίμα το ότι έφυγε ο κύριος Γκάιερ γιατί ήθελα πραγματικά να παραδεχτώ ότι έχει δίκιο. Αυτή τη στιγμή πέρα από την μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζουμε έχουμε μια δημοσιονομική ευκαιρία δηλαδή το ότι απροσδόκητα τουλάχιστον για αρκετούς από εμάς έχουμε 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Και θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Κομισιόν μήπως θα είχε νόημα τα λεφτά αυτά να μην ε, πάνε ως συνήθως ε, πίσω στα κράτη-μέλη αλλά τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος τους να γίνει αποθεματικό για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την τεράστια πρόκληση η οποία θα συνεχίσει να υφίσταται. Και είναι νομίζω μεγάλης ε, σημασίας το να μην πάρουμε λεφτά με τη σέσουλα και να τα ρίχνουμε από εδώ και από εκεί, αλλά χρειάζεται μια στρατηγική, ένα πολιτικό σχέδιο να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους ε, που έρχονται στην Ευρώπη, δεν έρχονται για τουρισμό, ε, είτε τους διώκουν είτε είναι άσχημα τα πράγματα. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι κάθε ανθρωπιστική βοήθεια χρειάζεται και ένα πλαίσιο να υπάρχει για να πιάσει τόπο. Υπάρχει διαφορά παραδείγματο χάρη. Ε, αν σκεφτούμε παραδείγματο χάρη το ότι στη Γερμανία ε, βλέπουμε ότι πρέπει να εξοδέψουμε και εξοδεύουμε 10.000 ευρώ τουλάχιστον ε, ανά πρόσφυγα ανά έτος και θα μπορούσαμε να φτιάξουμε στρατόπεδα προσφύγων ε, πιο κοντά στις περιοχές της κρίσης όπου με τα ίδια λεφτά θα βοηθούσαμε 20 για να μην πω και παραπάνω άτομα. Δηλαδή δεν έχει νόημα μόνο να δίνουμε λεφτά αλλά να τα χρησιμοποιήσουμε και πιο αποτελεσματικά και να έχουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για να μην ε, καταπολεμήσουμε το ζήτημα μόνο εδώ, αλλά πιο κοντά στην ουσία, εκεί που γεννιέται. Αν το καταφέρουμε αυτό, νομίζω πως θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε τον Ευρωπαίο πολίτη στα μάτια. Και στη χώρα μου, στη Γερμανία, η κατάσταση είναι εκρηκτική και πραγματικά δεν θα ήθελα να μεταφερθεί όλη αυτή η διάθεση και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν κατεπηγόντως ε, να δούμε σοβαρά αυτό το οποίο πρότεινα και από την άλλη και εμείς θα πρέπει να παρακαλέσουμε την Κομισιόν να κάνει τις απαραίτητες προβλέψεις τις ε, δημοσιονομικές ε, για να είναι έτοιμες αν τελικά διατεθούν αυτά τα χρήματα. Ευχαριστώ. Γκάρθια Σάμπαλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σύντομη Έλεγα πριν στον κύριο Ντεπρέ ότι ήμουν πολύ ικανοποιημένη από αυτή την διορθωτική επιστολή της Κομισιόν γιατί είναι στο μήκος κύματος των όσων ψήφισαμε στην Επιτροπή μας. Άρα ε, έτσι επομένω ε, συναντιέται η μία άποψη με την άλλη όσον αφορά την υποδοχή των προσφύγων και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Οπότε καλυπτόμαστε και άρα εντάξει, θα πρέπει να συζητήσουμε μετά της εγγύηση των νέων στον ε, ε, τριμερή διάλογο και το σχέδιο Γιούγκερ για το Euro Facility λοιπά. Αλλά ε, τα μισά τα έχουμε κάνει. Ο πάντως, αυτό το οποίο παρουσιάζει η Επιτροπή δεν είναι ακριβώς αυτό που εμείς ψηφίσαμε για τους πρόσφυγες και με ανησυχεί κάτι. Και αυτό δεν είναι σχόλιο. Κάτι σαν πρόταση προς την Επιτροπή είναι κάτι για τις ε, υπηρεσίες. Γιατί εμείς ψηφίσαμε αύξηση. Παραπάνω από την αύξηση που λέει τώρα η Επιτροπή για την ΕΑΣΟ Και είχαμε προτείνει επίσης και λιγότερη αύξηση από όσα λέει η Επιτροπή για την Frontex. Άρα πρέπει να λύσουμε το θέμα των υπηρεσιών γενικώ έχουμε για τον εισηγητή μας για τις ε, αποκεντρωμένες υπηρεσίες αλλά ενώ συμφωνούμε στις γενικές γραμμές δεν νομίζω ότι έτσι λύνεται το πρόβλημα των αποκεντρωμένων υπηρεσιών και ότι η ενίσχυση του ε, προσωπικού όπως προτείνεται θα βρει σύμφωνα τουλάχιστον την πολιτική ομάδα των σοσιαλδημοκρατών να ληφθεί υπόψη αυτό το οποίο ψηφίσαμε σας το λέω σαν πρόταση, σαν ε, ε, πρότασή μου. Όταν έρθει των διαπραγματεύσεων να το συζητήσουμε. Το συζητήσουμε και με το Συμβούλιο. Να ξέρετε ότι αυτό θα πρέπει να είναι στο τραπέζι. Μιλάμε για τον διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 8 και το θέμα του δισεκατομμυρίου ας το συζητήσουμε αργότερα. Δεν ζητάει άλλος κανείς το λόγο. Μόνο μία ερώτηση από μένα. Πολλής λόγος γίνεται για το ζήτημα της καταπολέμησης των αιτίων της μετανάστευσης. Διότι αυτό που προξενεί διαμαρτυρίες ή εκδηλώσεις αγανάκτησης τιμού είναι ο όγκος των ροών. Έχουμε διαρκώς την εντύπωση ότι αυξάνεται ο αριθμός. Μας το είπε και η κυρία Γεωργίου. Το αποτέλεσμα που θα θέλαμε να πετύχουμε δαπανώντας όλα αυτά τα ποτά είναι να πάψει η μετανάστευση. Οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων λοιπόν μιλήσαν για τη δημιουργία συνοριοφυλακής ή ακτοφυλακής Λαμβάνεται αυτό υπόψη στη διευθυντική επιστολή πέραν των τριών δις που μπορεί να αναφέρθηκαν. Κύριε Μαραγκάλη, νομίζω ότι η κυρία Μέρκελ είχε την εντολή ε, κατά κάποιο τρόπο από την κυρία Μογκερίνη που είναι, είπατε, εκπρόσωπος ε, για τις εξωτερικές υποθέσεις <clears throat> να παρουσιάσει αυτή την πρωτοβουλία, κάτι τέτοιο μάλλον συνέβη. Έτσι λοιπόν, εφόσον η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις ψηφοφορίες της Επιτροπής ε, Προπολογισμών, πέραν του Connecting Europe Facility και του Ορίζοντα 2020, το ιδανικό θα είναι να ακολουθήσει και το Συμβούλιο. Βέβαια θα πρέπει να αποφανθεί το Συμβούλιο στο σχέδιο επιστολής παριθμών 2 αλλά ίσως αυτές τις ερωτήσεις κύριε Φρέσκο, να μπορέσετε τώρα να τις απαντήσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις. Καταρχάς να τονίσω το γεγονός ότι πράγματι υπάρχει σύγκληση μεταξύ των όσων ψήφισε στις τροπολογίες της στο σχέδιο προπολογισμού 2016 αυτή η Επιτροπή, η δική σας, και όσων προτείνονται στη διευθυντική επιστολή υπαριθμών 2. Με διαφορετικό τρόπο ο κύριος Ντεπρέ, η κυρία Γκαρδιαθάμπαλ το είπαν. Φαίνεται να υπάρχει σύγκληση απόψεων σε πολλά θέματα. Τώρα για τις ερωτήσεις που τέθηκαν με τη σωστή σειρά. Ο κύριος Γκάγερ και ο κύριος Κόμινερ. Κέλμελ, ε, αναρωτήθηκε για το ρόλο της Frontex και όντως αν μου επιτρέπετε θα χρησιμοποιήσω τον αγγλικό όρο διότι ε, έχω την ορολογία πιο πρόχειρη στα αγγλικά από ότι στα γαλλικά για την περίπτωση των επιστροφών δεν υπάρχει θέμα πρωτοβουλίας για την ε, Frontex όμως συζητήθηκε το κατά πόσο η Frontex μπορεί να προβλέψει τα συνοδευτικά μέτρα για τις επιστροφές, να οργανώσει κοινέ πτήσεις για επιστροφές προς τις χώρες προέλευσης, για όσους έχουν τη αλλά δεν έχουν δικαίωμα να το λάβουν. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους όσο το δυνατόν περισσότερο. Ενώψη μια ενδεχόμενη αναθεώρηση ε, του των τη Frontex, όπω ανακοίνωσε ο πρόεδρο Γιούνκερ και όπω θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλο τη χρονιά, όντω χρειάζεται να ξαναδούμε εκ βάθρων το ρόλο τη Frontex και πώ διαφρώνεται με την δράση των κρατών μελών. Καθώ και την κυριαρχία του βεβαίω και τα δικά του δικαιώματα σε αυτήν. Αλλά εδώ χρειάζεται μια συλλογική απόκριση που να είναι αποτελεσματική δραστική και να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι μέρος της εξήγηση για τα επιπλέον μέσα που προτείνονται στον διευθυντικό προπολογισμό, στη διευθυντική επιστολή, Για τις υπόλοιπες πτυχές που αφορούν τα εσωτερικά μέτρα για την πρόκληση αυτή του μεταναστευτικού. κύριε Ντεπρέ, ρωτήσατε εάν στη διδοτική επιστολή συνδυάζουμε τα μέτρα αυτά με τη δεύτερη μέσμη. Ναι, 110 εκατομμύρια προστίθενται για το πρώτο πακέτο των 40.000 που πρέπει να επανακατασταθούν, ε, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών, των αντιπορικών που δεν ε, καλύπτονται αρχικά. Η αρχική πρόθεση λοιπόν είναι αυτά τα δύο να ευθυγραμμιστούν. Για την ονοματολογία τους τίτλους στον ε, τομέα των ετούντων άσυλων και των επιστροφών η δημοσιονομική διάρθρωση στους τελευταίους λογαριασμούς ε, της εκτέλεσης των ποσών απαιτεί κάποια ευελιξία ιδίως ως προς την ένταξη, στη συμπερίληψη ή τις Για τις επίγουσες λοιπόν τράσεις, αυτές που πρέπει να ολοκληρωθούν κατά επίγοντος, πρέπει να δούμε κατά πόσον καλύπτονται οι ανάγκες απόκρισης από την ονοματολογία που χρησιμοποιείται, από τους τίτλους που δίδονται στον προπολογισμό. Η λεπτομερέστερη κατανομή ε, απειλή να περιπλέξει περισσότερα τα πράγματα στην, στη φάση της υλοποίησης. Εδώ λοιπόν το λέω αυτό για λόγους ε, επιφυλακτικότητας από μέρους μας. Μα συγχωρείτε, εάν επιτρέπετε ο κύριος Ντεπρέ θέλω να σας διακόψει. Κύριε Ντεπρέ, ναι, κατανοώ την επιχειρηματολογία του κυρίου Φρέζα ε, και την σέβομαι πολύτως. Αυτό όμως που ρωτώ είναι αν αυτή η ειδική δημοσιονομική γραμμή μπορεί να χρησιμοποιείται. Στην ίδια μιλούμε για υλοποίηση μέτρων για την ένταξη και μέτρα για την επιστροφή. Δεν βλέπω πώς γίνεται να μεταφέρονται πιστώσεις από το ένα στο άλλο. Δεν βλέπω τη λογική. Ε, καταλαβαίνω ότι στις άλλες δημοσιονομικές γραμμές υπάρχει μια λογική μεταφορά των ε, ποσών. Όμως μου φαίνεται πραγματικά αξιοπερίεργο αυτό στη συγκεκριμένη δημοσιονομική γραμμή. Ε, κύριε Φέζα, έχετε το λόγο. προτείνω να συνεχίσουμε την ε, συζήτηση, διμερώς ίσως. Ίσως με τη βοήθεια των συναδέλφων που είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση. Μπορούμε να έχουμε έτσι και πιο ε, τεκμηριωμένες συζητήσεις. Ε, για τα υπόλοιπα θα τα ξαναδούμε μετά. Έχω σκοπό να απαντήσω γιατί τα έχω σημειώσει όλα κατά λεπτός. Κύριε Πρόεδρε, ρωτήσατε εάν η διορθωτική επιστολή προβλέπει μέτρα για Η συνοριοφυλακή στην Ευρώπη. Η απάντηση είναι όχι. Όχι στη διορθωτική επιστολή. Αυτή η ιδέα είναι όμως ε, αυτή τη στιγμή στο κέντρο των ε, ανησυχιών της Επιτροπής και σχετικές νομοθετικές προτάσεις θα γίνουν αρκετά σύντομα. Μα είναι καταπήγον οι προσελεύσεις καθημερινά, βλέπουμε τις εικόνες στην τηλεόραση, βλέπουμε πόσα άτομα έρχονται στα σύνορα και τα περνάνε. Δίκαιο έχετε, αλλά όλοι το καταλαβαίνουν αυτό πόσο κατεπήγον είναι, αλλά ταυτόχρονα αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τις πρόσφορες συνθήκε για να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία στο νομικό επίπεδο με το νομοθετικό πλαίσιο που διαθέτουμε. Υπήρξε έκκληση προ τη Frontex για να διατε... από τη Frontex μάλλον, για τη διάθεση εμπειρογνωμόνων από τα κράτη-μέλη για όσους έχουν τις ειδικές γνώσεις και δυνατότητα και προκειμένου να υπάρξει άμεσα καλύτερο έλεγχο στα σύνορα, σε αυτή τη μεταβατική φάση υπάρχουν και δράσει που διεξάγονται για να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στι ανάγκε αυτέ τη μεταναστευτική πίεση. ως προς το ρόλο των οργανισμών και την ενδεχόμενη ενίσχυσή τους σημειώνω σε κυρία Γκαντία Θάμπαλ ότι πρέπει να δούμε με μεγάλη προσοχή την κατάσταση των οργανισμών και βεβαίως αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν στις διαπραγματεύσεις. Είτε ξεχωριστά, είτε προληπτικά όπως προτείνει ο κ. Γκάιερ, αλλά βεβαίως εδώ θέλουμε να συμπαραταχθεί μαζί μας και το Συμβούλιο ή να το πείσουμε στη συγκελαγή Για τα τρία δις για την Τουρκία. Να υπογραμμίσω ότι αυτά τα τρία δις είναι μεταξύ μεγέθους που προηγουμένως συζητήθηκε. Δεν ήταν συμπέρασμα το οποίο κατέληξαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σκοπός ήταν να ενισχυθεί η συνεργασία με την Τουρκία που είναι παράγοντας κλειδί στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. στιγμή αυτό που έχει ήδη καταστεί σαφές είναι το, το καταπίστευμα για την ε, Συρία, το λεγόμενο μαντάτ που θα πει ελπίδα στα αραβικά, φτάνει κατά ε, τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 500 εκατομμύρια. Θα διορθωθεί αυτό το ποσό από την γραμμή του προγράμματος του προενταξιακού, του ΕΜΠΑ. Εδώ σκοπός είναι να υπάρξει αντιστοίχηση από την πλευρά των 100 μελών και να υπάρξει απαραίτητη κρίσιμη μάζα για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Αυτό το καταπίστευμα θα είναι το βασικό μας όχημα και εδώ θα χρειαστούμε τους πόρους του ευρωπαϊκού προπολογισμού αλλά και τις συνεισφορές των κρατών μελών στον ίδιο βαθμό. Ο... Έτσι ορίστηκαν τα τρία δις κατά τις διαπραγματεύσεις και ο... έτσι θα έχουν ε, εγκριθεί εφόσον ολοκληρωθούν. Θα φανεί τις ερχόμενες εβδομάδες. Για τα γεωργικά. Ο κύριος Τόρβαλτ μίλησε κυρίως μίλησε κυρίως για το χείριο εδώ στη διευθυντική επιστολή 29 εκατομμύρια προβλέπονται για το χείριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά. Εάν χρειαστεί, θα υπάρξει δυνατότητα να απαντήσουμε καταλήλως. Απλώς να θυμίσω, ίσως το θυμάστε, τα συζητήσαμε και πριν ένα χρόνο, με την απόκριση στο ρωσικό εμπάρκο. Τότε με διαδοτική της επιστολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει διόρθωση στις δαπάνες Η ερώτηση τότε ήταν αν είναι επαρκής και αν η χρήση του αποθεματικού για τις κρίσεις γίνονταν σωστά. Ένα χρόνο μετά μπορούμε να πούμε πως ναι. Οι αναλήψεις πιστώσεων ήταν αρκετές όπως είχαν προβλεφθεί και τελικά είχαμε και σωστή υλοποίηση ένα χρόνο μετά. Οπότε να θυμίσω ότι προσέχει πάρα πολύ την πρόληψη των αναγκών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τα διαφορετικά είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί η κατάσταση βάσει των όσων ξέρουμε εκ των υστέρων. Ελπίζω να μην ξέχασα πολλέ ερωτήσει, αλλά εφόσον χρειαστεί μπορώ να επανέλθω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Φρέζα. Αναφέρθηκε η Frontex. Αλλά κάποια από τα μέλη τη Επιτροπή εδώ είχαμε πάει τον Ιούλιο στην Σικελία και θα ενημερώσουμε από κοινού του συναδέλφου τη Επιτροπή ΛΥΜΠ και του συναδέλφου εδώ για τα όσα είδαμε εκεί. Υπήρχε δυσφορία στη Σικελία. Αναρωτιόνταν τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνουν οι οργανισμοί τη. Έχουμε την εντύπωση ότι κρατάει στατιστικά αρχεία η Frontex. καταγράφει το πόσοι υπέρασαν παράνομα τα σύνορα, αλλά σαν παρατηρητή. Δεν υπάρχει πραγματική δράση. Όλες οι πρωτοβουλίες παραμένουν στα χέρια των κατωμελών. Και αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Εάν ο ρόλος της Frontex ενισχυθεί, θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Αυτό που μας ανησυχεί είναι να δούμε πώς θα δίνονται οι εντολές από ένα κεντρικό επίπεδο. Πού θα βρίσκεται η κυβέρνηση, δηλαδή αυτή η εξουσία που θα μπορεί να κυρώνει τις αποφάσεις. Αυτά θα τα ξανασυζητήσουμε, αλλά επειδή αυτή η κρίση είναι ανευπροηγουμένου, και τώρα βρισκόμαστε μόνο στις αρχές της, νομίζω ότι μπορεί, μπορεί κανείς να εκφράσει ενδιασμούς, ενδιασμούς για την δημοσιονομική απόκριση που προβλέπετε, έτσι όπως διαφαίνεται τουλάχιστον. Και ακόμη και αν η διευθυντική επιστολή υπαριθμού 2 αποτελεί ένα πούμε πρόοδου, είμαι βέβαιο ότι θα χρειαστούμε έκτακτα μέσα, εάν θέλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνε μας το 2016. Προδήλως σήμερα δεν το έχουμε καταφέρει αυτό. Και αναρωτιέμαι εάν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έχουν πραγματικά ε, σταθμίσει σωστά το τι συμβαίνει. Τούτων λεχθέντων θα περάσουμε ε, τα επόμενα θέματα, καθότι η διδοτική επιστολή μας φαίνεται ελπιδοφόρα, αλλά αυτό θα μας πούν δεν μας αφορά και καθότι η ε, κατανομή του προπολογισμού σωστά είναι ένα όνειρο που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στι σχέσει μεταξύ των κατομελών. ΤΕΠΟ και ο κ. Ντεπρέ σωστά και εσεί κύριε Φρεζά θα μα επιτρέψετε να είμαστε ακόμα γεμάτοι ελπίδα σε ένα βαθμό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα περιγράψω τα στοιχεία του διορθωτικού προπολογισμού περιθμών 8. Λοιπόν, πρόκειται για στατικό προπολογισμό, τόσο ώστε να μπορέσουμε να επικαιροποιήσουμε αυτή την ε, βάση υπολογισμού των ιδίων πόρων. Και έτσι καθορίζεται ε, το πόσο θα πρέπει να καταβάλουν τα κράτη-μέλη για τον προπολογισμό. Και φέτος, ο τροπικό προπολογισμό έχει τρεις άξονες βασικά. Πρώτα-πρώτα, από πλευρά επιπτώσεων είναι το πιο σημαντικό, κάτι σαν ανακύκλωση κάποιων εκκρεμών από πέρσι. Θυμάστε ότι είχε χρειαστεί κάποια ρύθμιση για τη χρήση του 2014 όσον αφορά τον ΦΠΑ και το ΑΕΠ. Επίσης έχουμε κάποιες πληρωμές έξι κρατών μελών. Οι χώρες αυτές ανέβαλαν κάποιες πληρωμές του 2015 και την 1η έγιναν αυτές οι περίμερες πληρωμές από τα κράτη-μέλη και αυτά όλα αντιστοιχούν σε ποσό 5,7 δις που πρόκειται να αναδιανεμηθούν για όλα τα κράτη-μέλη. Ο δεύτερος άξονας τώρα είναι κάτι πάγια υπάρχει είναι ότι πρέπει να δούμε τις ε, ε, αναθεωρημένες ε, ισορροπίες για το ΦΠΑ και το ΑΕΠ οπότε και έχουμε και αναθεώρηση των προγνώσεων για τις συμβολές που θα πρέπει να τα κράτη-μέλη. Και αυτό το στοιχείο αντιστοιχεί σε 1,4 δις για όλα τα κράτη-μέλη. Το τρίτο στοιχείο, σημαντικό και αυτό, είναι το ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα επιπλέον έσοδα από τελωνιακούς δασμούς. Πρόκειται για πρόστιμα από την πολιτική ανταγωνισμού. Και αυτή η τελωνιακή δασμή είναι 0,8 δις περισσότερο από όσα αρχικά είχαν εγγραφεί στον προπολογισμό. Πρόκειται κυρίω για τόκους και πρόστιμα. Και φτάνουμε στο 1,5 δις περισσότερο από όσο είχε εγγραφεί και προϋπολογιστεί. Επίσης είπαμε ότι στον διορθωτικό υπαριθμόν 8 υπάρχουν και προβλέψεις για την ε, υπηρεσία προστασίας των δεδομένων και μείωση δαπανών κατά κανόνα 3.000 ευρώ. Να και να τώρα τα έσοδα και να δούμε τι είπε ο κύριος ε, Γκάι ο κύριος Κόλμα. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το διακύβευμα. Είναι θέμα, αν θέλετε, Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή, τον εξεταστούν οι διάφορες πηγές ε, εισοδήματος και εσόδων και πρέπει να γίνουν σχετικές προσαρμογές. Αυτό όμως δεν έχει άμεσες επιπτώσεις όσον αφορά τις ε, πιστώσεις σε σχέση με τις δαπάνες που έχουν προϋπολογιστεί γιατί το σύστημα μας το δημοσιονομικό προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται κάποια έγκριση όσον αφορά τις υποχρεώσεις και όσον αφορά τις ε, πληρωμές για τις δαπάνες. Ε, όριο και περιορισμός είναι οι οροφές του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και επί τη βάση των ε, δαπανών που έχουν γραφεί στον προϋπολογισμό υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πόσοι ήδη πόροι θα πρέπει να εισπραχθούν από τα κράτη-μέλη. Και μέσα στη χρονιά γίνεται αναθεώρηση αυτών των ε, υπολογισμών και λαμβάνεται υπόψη η ίσπραξη των τελειωνικών εγκοντασμών τι γίνεται από πλευράς ΦΠΑ και ΑΕΠ και έτσι κάνουμε την προσαρμογή των ε, εσόδων. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε 9,4 δις περισσότερο από τα κρατημέλια. Όμως αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι έχουμε περισσότερα έσοδα από τους δασμούς και από το πρόστιμα. Κάτι που δεν είχε προϋπολογιστεί. Και ε, έχουμε είπαμε σύνολο 2,3 δις και αυτό αντιστοιχεί αναλογικά με το ΑΕΠ σε όλα τα μελη Οπότε έχουμε κατανομή στα ΑΕΠ στα κράτη-μέλη συγγνώμη, του βάρους της χρηματοδότησης του προπολογισμού. Δεν ωφελούνται όλοι το ίδιο. Ε, υπάρχουν προσαρμογές, κάποιοι πρέπει να συμβάλλουν περισσότερο, κάποιοι λιγότερο. Ανάλογα με αυτές τις ε, προσαρμογές του υπολογισμού των ιδίων πόρων. Τώρα, γιατί δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα κονδύλια η Επιτροπή, τα, τα πρόστιμα και τους ε, δασμούς. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει η έγκριση για αυτές τις πιστώσεις. Δεν είχε συμφωνηθεί στον Πολιτισμό και έτσι για να αυξηθεί η δαπάνη το Συμβούλιο πρέπει να συμφωνήσει με το Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω, ας πούμε, στο κεφάλαιο 2 ή 3. Και έτσι, σύμφωνα με τους κείμενους κανόνες, υπολογίζονται οι διπόροι. Και αυτό καθορίζει το πόσα θα συνεισφέρουν τα κρατημέλη. Και όταν τέλος της χρονιάς έχουμε 2,3 δις από αυτά τα έσοδα που είναι παραπάνω από όσα είχαν στην αρχή ε, προβλεφθεί, αυτό δεν πάει να πει ότι πρέπει, μπορεί η Κομισιόν να δαπανίσει περισσότερο. Για να δαπανίσει περισσότερο θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από τις δύο ε, αρχές του προπολογισμού. Δυστυχώ επομένω δεν προβλέπεται τέτοιου είδου ανακύκλωση, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Α, ωραία, επομένω πάει το όνειρο αυτό και επανερχόμαστε στην πραγματικότητα την δημοσιονομική. Κυρία Γενική Συντηρία η συγκήτρια, συγγνώμη, για το 2015. Ναι, ευχαριστώ. Κάθε φορά που έχουμε διορθωτικό προπολογισμό που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, διαπιστώνουμε ότι πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουν οι αυτά τα χρήματα που πρέπει να πάνε πίσω στα κράτη-μέλη. Για αλήθεια είναι ότι, ότι πολλές φορές πέφτουμε σε παγίδε. γιατί όπω είπε η Κομισιόν έχουμε αυτό το 1 δισεκατομμύριο. Είναι θέμα ε, προπολογισμού. Δεν μπορούμε να τα ξοδέψουμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, και ακόμα και να το κάνουμε αυτό θα είναι άσχετο με τα 9 δι. Τέλος πάντων θα χρειαζόταν να αυξηθεί η οροφή, να κάνουμε μια κατεπίγουσα διόρθωση να το δοκιμάσουμε. Αλλά θα ήταν μπλεγμένο. Νομίζω ότι όσον αφορά το δημοσιακό πλαίσιο να μείνουμε εκεί που από το 2016 και να βαδίσουμε με λογική και νυφαλιότητα. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχουμε αυτά τα 9 δις και είπαμε ότι έχουμε δύο δις που δεν είχαν προϋπολογιστεί και προέρχονται από τα πρόστιμα κλπ. Ε, υποθέτω ότι αυτό σίγουρα θα διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ε, καλύτερα περισσότερα παρά λιγότερα για το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα αλλάζουν τα πράγματα και για αυτούς που θα έρθουν να διαπραγματευτούν μαζί μας. Άρα κάτι καλό είναι αυτό για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Πάντως, Ούτε τεχνικά ούτε νομικά δεν γίνεται, αλλά πολιτικά γίνεται. Μπορούμε να προτείνουμε στο Συμβουλίο ότι μια και έχουμε αυτά τα έξτρα χρήματα, θα μπορούσαμε ας πούμε αυτά τα οποία εισπράχθηκαν από τα πρόστιμα να αξιοποιηθούν από τα 28 κράτη-μέλη. και έτσι τα κρατημέλη να εισφέρουν όπως οφείλουν για αυτό το καταπιστεύμα για τη Συρία. Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι αν θυμάμαι καλά έχουμε εκείνο το πρόγραμμα της εμπιστευτικής βοήθειας και δεν είχε καλυφθεί η διεθνής βοήθεια που είχε προβλεφθεί και να πούμε στο Συμβούλιο ότι όχι ως όργανο αλλά η κάθε χώρα χωριστά να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πόρους ούτως ώστε να καλυφθούν τα κενά του προγράμματος του επισητιστικού ούνρα κλπ. Οπότε μπορεί να μην ε, ε, είναι να η δαπάνη με άλλο τρόπο, αλλά μπορούμε να προτείνουμε κάτι τέτοιο και να ελπίζουμε ότι θα είναι θετική στάση του Συμβουλίου. Αυτό και έγινε από την ε, γενική μας συγκέντρια. Το ερώτημα είναι από πού θα εμφανιστούν αυτές οι επιστώσεις. Στον προπολογισμό της Ένωσης θα εμφανιστούν στις δημοσιονομικές γραμμές των κρατών μελών, στους εθνικούς προπολογισμούς δηλαδή, στα επίπεδο των Υπουργείων Οικονομικών. Όταν μιλάμε για συνεισφορές που ε, περνούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, αυτά τα δύο δις σίγουρα δεν θα πάνε χαμένα, θα επιστρέψουν στα κρατημέρια. Εάν βάλω το χέρι στην τσέπη τα κάτι μέλη για να, για να καλύψουν τα τρία δεκαδείς και για να υπάρξει συνοροφυλακή και εκτοφυλακή κάπου θα πρέπει να βρούμε αυτά τα χρήματα. Και όπως ο δυναμικός κανόνας ε, προβλέπει ότι οι δαπάνες δεν αντιστοιχούν, ε, πρέπει να αντιστοιχούν κανονικά στα έσοδα, θα πρέπει να βγουν από κάπου αυτά τα τρία δις. Σε ό,τι αφορά τι μεταναστευτικέ πολιτικέ, και σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό της Ένωσης. Αυτό είναι ένα πράγμα και άλλο οι άμεσες ανασφορές, τα ποσά που άμεσα εκταμιεύουν τα κράτη-μέλη προς, την, προς τον ΟΗΕ ή προς κάποια τρίτη χώρα, την Τουρκία, την Ιορδανία, το Λίβανο. Νομίζω ότι θα παραμείνουμε σε αυτά, διότι η κατανομή των πόρων αυτή τη στιγμή σε έκτακτες συνθήκες μας παραπέμπει στην τόσο ε, δυσχερή και τόσο ματαιωτική η διαδικασία συναλλαγή που θα ακολουθήσει, αλλά αυτό κάπως μα ανανεώνει ε, αναγκαστικά. Κύριε Μαραγκάλ, πολύ σύντομα να συμφωνήσω απολύτω με αυτά που είπε η κυρία Γκαρδιά Θάμπαλ και να προσθέσω κι εγώ ένα στοιχείο παραπάνω. que hoy tenemos encima la mesa es que este Parlamento está en condiciones de ser. Να του πούμε ότι το Κοινοβούλιο κατηγορηματικά και απόλυτα θέλει να προστατεύσει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων και ότι στις επαφές και διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο εκεί υπάρχει ένα στοιχείο ιστορικό το τι γίνεται με τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Και επομένως ότι υπάρχει τώρα το περιθώριο να κάνει η Ευρώπη αυτό το οποίο πρέπει. Επομένως αυτή θα πρέπει να είναι η αφετηρία. Αυτό το οποίο εμείς θα απαιτήσουμε. Δηλαδή να λάβουμε υπόψη αυτό που επιτάσσει πραγματικότητα. Merci. Il n'y a pas d'autres demandes de parole. Je pense que Ευχαριστώ. Δεν ζητάει άλλο κανεί το λόγο. Καλό θα ήταν λοιπόν σύντομα να έχουμε μια ανακεφαλαίωση, να δούμε ακριβώ πώ θα διαμορφωθεί η μεταναστευτική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάποια στιγμή για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών να ξέρουμε τι θα περνάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη και ποιε θα είναι οι άμεσε συνεισφορέ των κρατών μελών. Το έγγραφο λοιπόν που θα τα καταγράφει όλα αυτά ε, βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας. Έτσι κι θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε στο επίπεδο της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάτι να προσθέσει, αν και έχω την εντύπωση ότι όλα τα καλύψαμε, τα καλύψαμε όλα μάλλον σε σχέση με το θέμα. Ε, καλωσορίζω εδώ τον κύριο Λάρσεν που είναι διευθυντής προσωπικού και τον κύριο Σεφ που είναι διευθυντής για την ε, Αμερικανική Ήπειρο την έδ και θα σας ενημερώσω για τη δικασία πρόσληψης ενός ειδικού συμβούλου ε, για τα θέματα της Κολομβίας. Ο ποιος θέλει το λόγο, ο κύριος ε, Λάρσον ή ο κύριος Σέπφερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λάρσον, λέγομαι. Ναι, πράγματι. Η ύπατη εκπρόσωπο σκοπεύει να ορίσει ειδικό απεσταλμένο τον κύριο Γκίλμορ, πρώην Υπουργό Εξωτερικών τη Ιρλανδία, τον κύριο Πετρέιτ, πρώην Αντιπρόεδρο τη Κυβερνήσεω, ω ειδικού συμβούλου με ε, καθήκον την ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία ε, προς όφελος της ειρήνης εκεί πέρα και για τον συντονισμό της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία. Αντιλαμβάνω πως κυρίως σας ενδιαφέρει η αμοιβή βεβαίως των απεσταλμένων, οπότε θα σας αναφέρω τις λεπτομέρειες. Θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο, 1η Νοεμβρίου, και θα συνεχίσει να εργάζεται από την Ιρλανδία. Με αποστολές βεβαίως. Αλλά με βάση την Ιρλανδία. Επίσης ε, δεν θεωρούμε ότι πρόκειται για δουλειά πλήρους απασχόλησης. Υπολογίζουμε ότι θα απασχολείται κάθε δύο εβδομάδες ανά δύο μήνες ε, με διάρκεια σύμβασης ένα έτος. 84 ημέρες εργάσιμες δηλαδή και θα αμυφθεί επίσης και με per με ένα 22ο του βασικού μισθού ενός ε, υπαλλήλου με βαθμό AD16 που του αντιστοιχεί και εάν ε, είναι όντως αυτός ο φόρτος της εργασίας μιλάμε για μια ετήσια αμοιβή 50.000 ευρώ. Θα καλύπτονται βεβαίως τα έξοδα των αποστολών από την υπηρεσία μας, όμως δεν θα έχει κάποια άλλη γραμματιακή υποστήριξη ή τίποτα άλλο. Θα βασίζεται στην υπηρεσία μας, είτε στις Βρυξέλλες είτε στις αντιπροσωπείες. Και βεβαίως θα πρέπει να δηλώνει όλες τις άλλες δραστηριότητες του κτλ. Αυτά εν ολίγης έχουμε προβλέψει. Κύριε Γκυλμό, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ντεπρέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μόλις άκουσα τον εκπρόσωπο της ΕΕΔ και είπε ότι είμαστε αρμόδιοι για τις αμοιβές. Όντως, μεταξύ των αρμοδιοτήτων έχουμε περιορισμό μέχρι τις αμοιβέ. Αλλά πρέπει να δούμε κατά πόσο οι αμοιβέ είναι έπλογε και κατά πόσο η αποστολή που ανατίθεται είναι εύλογη. Για το... Για το κόστος λοιπόν δεν μπορώ να κάνω ε, σχόλιο. Απλώ αναρωτιέμαι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από αντιπροσωπεία στην Ποκοτά. Η αντιπροσωπεία αυτή είναι σε θέση να κάνει τις σωστές ε, διαδικασίε σωστού συνδυασμού της ερευνητικής διαδικασίας στην Κολομβία και των όσων συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδαλώ δεν έχει νόημα. Θέλουμε να καταλάβουμε ποιο είναι ο χαρακτήρα τη προστιθέμενη αξία, τη παρουσία αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση επί τόπου και αυτού του ειδικού του επιτετραμένου μάλλον. Ε, επίσης, καταλαβαίνω γιατί μπορούμε να αποστείλουμε έναν επιτετραμένο αν μια από τις δύο πλευρές, αλλά δεν υπόθηκε αυτό, εφόσον ισχύει έχει καλός, αλλά δεν υπόθηκε, εάν στην ειρηνευτική διαδικασία συμμετέχει μια από τις δύο πλευρές και έχει εκφραστεί επιθυμία για την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συμμετέχει στη δικασία σχέση στις ε, διαπραγματεύσει. Υπάρχουν σχετικά έγγραφα, ε, υπάρχουν μαρτυρίες ή μια πραγματική επιθυμία ως προς αυτό και μια γενικότερη σκέψη. Υπάρχουν πολλοί επιτετραμένοι που είναι πρώην υπουργοί, πρώην επίτροποι και έχουν διαφορετικές ε, και ποικίλε αποστολές. Αυτό παρατηρώ και διερωτώ με. Είναι ένας από τους ρόλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για μερικούς ανθρώπους που σίγουρα είναι εξαίρετες προσωπικότητες αλλά των οποίων οι αρμοδιότητες που ανατίθενται συνήθως δεν δικαιολογούνται από την πραγματικότητα. Μιλάτε για ένα Κύριε Τζάνι, ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να προσθέσω μια-δυο ερωτήσεις σε αυτές τις πολύ συγκεκριμένε που έθεσε ο κύριος Ντεπρέ και με τις οποίες συμφωνώ. Ξεκινώ από το γεγονός ότι όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είμαστε υπεύθυνοι και για τις αμοιβέ. Δεν είμαστε μάλλον ακριβώ υπεύθυνοι για τι αμοιβέ, αλλά κυρίως για το κατά πόσον είναι εύλογες ε, τα άτομα τα οποία αναλαμβάνουν μια, μια θέση, κατά πόσο είναι προετοιμασμένοι και επί της ουσίας έχουν τις γνώσεις για να το αποκριθούν. Οι ερωτήσεις μου είναι τέσσερις. Η πρώτη αφορά το πόσα άτομα απασχολεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη στην Κολομβία και εδώ για τις σχέσεις με τη χώρα αυτή. Καλό θα ήταν για να το καταλάβουμε σε σχέση με το τι πόροι ήδη διατίθενται. Έπειτα, εάν η Επιτροπή μπορούσε να διευκρινίσει τι αρμοδιότητες θα έχει αυτός ο ειδικό σύμβουλος. Διότι στην εισαγωγή ήταν αρκετά γενική η εικόνα, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες. Γιατί αυτή την περίοδο δεν θα είναι στην Κολομβία αλλά από κατάλαβα θα δουλεύει κυρίως από την Ιρλανδία και θα μετακινείται απλώς εφόσον χρειάζεται για ορισμένες αποστολές στην Κολομβία. Και σε τι φάση βρίσκεται η ειρηνευτική διαδικασία. Δεν έχω εμβαθύνει. Ε, Στι συνεδρίε των συντονιστών για το σημείο αυτό εκφράστηκαν πολύ για την ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία και για το κατά πόσον έχει προχωρήσει αρκετά ή ε, κατά πόσον η πορεία έχει τόσο πολύ προχωρήσει που να δικαιολογείται και παρουσία εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, συμφωνώ δηλαδή εδώ με την ερώτηση του κυρίου Ντεπρέ. Θα πρέπει να υπάρξει έκφραση επιθυμίας από μια από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές για την παρουσία τρίτου παρατηρητή συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέταρτη ερώτηση, ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες του πρώην Υπουργού της Ιρλανδίας για την Κολομβία. Ποιες θα είναι οι ιδιαίτερες γνώσεις και η συνεισφορά του. Δεν είναι σαφές ακόμα αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Έχω εγώ μια συμπληρωματική ερώτηση. Όλοι γνωρίζουμε εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πραγματική πολιτική εξωτερική, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν ε, την ε, τάση να διατηρούν και τη δική τους αυτόνομη εξωτερική πολιτική. Πέραν της εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κολομβία, μπορείτε να μα διαφωτίσετε για το κατά πόσο είναι παρούσε άλλε αντιπροσωπείε των υπόλοιπων ε, των 100 μελών μάλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, πώ συντονίζονται όλα αυτά. Πώς ε, γίνεται η θυγμάτιση των ε, ανθρωπίνων πόρων εκεί, αφόσον όλοι επιδιώκουν και την εξοικονόμηση. Μπορούμε να κάνουμε οικονομίες μένοντας τον αριθμό των μελών της αντιπροσωπείας και γεννέμοντας πιο σωστά, εξισορροπώντας τα μέσα. Θα μου πείτε άλλο οι αμοιβέ του επιτετραμένου, όμως ε, ως Επιτροπή Προπολογισμών θέλουμε να το καταλάβουμε και αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις, αν και κάπως ε, φεύγουν τις μου, αρμοδιότητάς μου, γι' αυτό θα δώσω τον λόγο στον κύριο Σεβερίν σε λίγο. Πρώτα απ' όλα, Μόλις ανέφερα το άρθρο 123 και την ε, προφορική πρόσκληση ε, όσον αφορά δηλαδή τις ε, συμβατικές υποχρεώσεις που προτείνονται γι' αυτό έμεινα σε αυτό και ελπίζω να ήταν σαφές και να σας έχουν κοινοποιηθεί αυτά. Ναι, έχουμε αντιπροσωπεία στην Πογκοτά για να απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. Δεν έχω τώρα πρόχειρα τα στοιχεία, πόσοι άνθρωποι δηλαδή ασχολούνται με την Κολομβία συνολικά και στην αντιπροσωπεία και στις Βρυξέλλες. Οπωσδήποτε μπορώ να σας τα δώσω τα στοιχεία. Γεγονός είναι πως είναι κάπως στοχευμένη η επιχείρηση, η λειτουργία εκεί πέρα, ασχολείται με μία πτυχή Ε, ανέφερα αποστολές ε, δεν θα είναι μόνο μεταξύ Ιρλανδίας και Κολομβίας, μπορεί να είναι και άλλες. Ε, δεν θα είναι επίσης μόνο στην αντιπροσωπεία στην Πογκοτά. Κάποιος ανέφερε ότι έχουν παραγίνει, έχουμε πάρα πολλούς ειδικού αποσταλμένους. Όχι! Όχι ιδιαίτερα. Εντάξει, δεν ξέρω για την Κομισιόν, αλλά αυτό είναι ο τρίτος μόνο που έχει η υπηρεσία μας. Έχουμε έναν για πειθαρχικά ζητήματα με την ίδια αμοιβή. Έχουμε έναν μη αμοιβόμενο για το θέμα του Ιράν, την κυρία Άστον, για να συνεχίσει να ασχολείται με το ζήτημα αυτό, την Βαρόνη Άστον, ε, και ο τρίτος για την Κολομπία, δεν είναι πάρα πολύ. Τώρα, για την αιτιολόγηση των πόρων το ανέφερα. Ε, για το δικό σας σχόλιο, κύριε Πρόεδρε. Οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο με απασχολεί πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις αντιπροσωπείες που έχουμε σε 140 σημεία. Το έχουμε ξεκινήσει αυτό και θα χρειαστούν πολλές ε, δεκαετίες ε, μέχρι να υπάρξει ένα σοβαρό σύστημα, αλλά υπάρχει οπωσδήποτε ενδιαφέρον των κρατών μελών να συνεργαστούν πιο στενά. Έχουμε πλέον ε, και συστέγαση, αλλά και δεδομένη της κατάστασης των προπολογισμών πολλών κρατών, λαμβάνουμε προτάσεις, μήπως μπορούμε να στείλουμε ένα διπλωμάτι μας σε εσά, στα γραφεία σας και τέτοια. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και είμαστε μόνο στην αρχή. Και ναι, ελπίζω να συνεχιστεί και οπωσδήποτε μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά θα δώσω τον λόγο στον συνάδελφο, κύριο Σεβερένη, αν μου επιτρέπετε, για την πολιτική πτυχή. Σας ευχαριστώ κύριε Λάρσον, αλλά Ωραία, τότε να κανονίσουμε ραντεβού και να τα πούμε. Αυτό για την ε, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αυτές τις μετακινήσεις, για αυτές τις ε, αποστολές όπως την Ουκρανία. Με αυτό δεν είναι αυτονόητο γιατί έχουμε εκπρόσωπο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οπότε ποιος έχει το πάνω χέρι δεν είναι σαφές. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Πέραν αυτόν τώρα για τα κυριότερα πολιτικά ζητήματα. Τι λέτε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αλλά θα είμαι σύντομος γιατί ε, έχουμε αυτές τις ε, ερωτήσεις οι οποίες ε, τελικά απόκεινται στην κρίση του πρόεδρου της Κολομβίας για το πώς έχει οριμάσει η διαδικασία της ειρήνευσης και σας διευκρινίζω ότι σε επαφή με την είπατε εκπρόσωπο είπε ότι θα ήθελε να υπάρχει εκπρόσωπος ε, του προσωπικού και να ε, πλαισιωθεί έτσι η διαδικασία της ειρήνευσης από και συναυθεί η συμφωνία άλλωστε τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει πολλά βήματα πρόοδου και επομένως ελπίζουμε ότι θα υπάρχει κάποιο είδους ε, χρονοδιάγραμμα λογικό και να καταλήξουμε εκεί που θέλουμε. Οπότε, να, τη ζήτησε από την κυρία Μογκερίνη ο πρόεδρος Σάντο. Merci, Monsieur est Est-ce que votre réponse appelle des questions, Monsieur Depré Ερωτήσεις, Depré De nous être donné. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση, γιατί είπαμε ότι ανταποκρινόμαστε σε κάτι που ζητήθηκε. Αυτό είπαμε. Βεβαίω και εξορισμού εμπιστευόμαστε την υπατική αλλά θα πρέπει στο φάκελο να διευκρινιστεί ότι αυτό έγινε αιτήση των Κολομβιανών αρχών που ζητήθηκε η παρουσία του ειδικού, της ειδικού εκπροσώπου. Ότι δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένη αποστολή με συγκεκριμένες συνέπειες στα πλαίσια αυτών των πολιτικών διπλωματικών επαφών. Οπότε με μεγάλη μου χαρά μαθαίνω ότι όλα αυτά ακολούθησαν αυτές τις επαφές, αυτή, αυτό το αίτημα του Κολομβιανού Πρόεδρου. Α, άκουσα γιατί τι είναι τον κύριο Γκίλμορ. Έχει και άλλες υποχρεώσεις. Τι θα κάνει, θα πάει στην Κολομβία, υπάρχει άλλη αποστολή. Τι λέτε. Είναι μια αποστολή που έχει πολλέ διαστάσει, πολλέ πτυχέ, αλλά και πολύ συγκεκριμένη. Πολύ καλά λέει ο πρόεδρο. Κύριε Ντεπρέ, είναι σαφέ. Δεν ήταν σαφέ, αλλά γίνεται κάπω πιο σαφέ από πριν. Άλλε ερωτήσει. Σα ευχαριστώ, οπότε μπορεί η Επιτροπή μας να ε, αποφανθεί χωρίς επιφυλάξεις. Και τώρα, Δοκιμάστε τις κάρτες σας στα μηχανήματα. Τι ώρα προβλέπονταν στις 11. 11.30. Mm. Θα πρέπει να διακόψουμε τη συνεδρίαση. Να την διακόψουμε. Je Σας επιβεβαιώνω ότι θα έχουμε συνεδρίαση στις 27 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο στις 14 και 15, 2 και 4 με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ε, κοινή συνεδρίαση. Το είπα, αλλά το βεβαιώνω, διότι τώρα ξέρουμε ότι έχουμε και την αίθουσα. Και θα έχουμε και υπηρεσίε διερμηνία, μετάφραση, λέει ο Πρόεδρο. Alors, notre, rapporteur général propose de voter maintenant. Θέλετε να ψηφίσουμε τώρα, έτσι προτείνετε κυρία Συγγήτρια. νόμιζα ότι υπήρχε θέμα παρουσίας βουλευτών, αλλά φαίνεται ότι είμαστε, έχουμε την απαραίτητη επαρτία για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Εντάξει λοιπόν, τότε να ψηφίσουμε τώρα. Οι συνάδελφοι που θα έρθουν στις 11.30 βέβαια μπορεί να μας... Ε, μπορεί να μας ε, το επισημάνουν αυτό και να μας προσέξουν. Αλλά θα πρέπει να ψηφίσουμε και για την αντικατάσταση συνεργάτη του κ. Μπούζεκ. Συνεχίζουμε λοιπόν τις εργασίες μας εκεί όπου είχαμε σταματήσει να δώσω το λόγο στην Έιντερ Καρδιαθάμπαλ για τις αιτήσεις μεταφοράς 30. Πρόεδρε, δεν υπάρχει εδώ πρόβλημα, απλώς έχουμε τη χρηστή 20.000 ευρώ που δεν έχουν δαπανηθεί για να βελτιώσουμε τα όσα έχουν γίνει τώρα, ως τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Προτείνω να υπερψηφίσουμε. Κάποιοι δεν θέλουν να ψηφίσουν. 13, 13 ε, κάρτες έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλά μόνο 11 ψήφισαν. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 12, 9 ε, ψήφους υπέρ, μία κατά και δύο αποχές. Και τώρα ο λόγος για τα λοιπά τμήματα. Ο κύριος Ντεπρέ που εκπροσωπεί την κυρία Χολμάγερ. Μα του έχει παραχωρήσει αυτή την αρμοδιότητα. Πραγματικά εξεπλάγεται από τότε αντιδράσεις ε, προξενή μεταξύ κάποιων από τους πιο συμπαθείς συναδέλφους, θα πρέπει να μας το εξηγήσουν ίσως. Υπάρχουν τρει τρεις προτάσεις μεταφορών που μας έχουν υποβληθεί και τις οποίες μελέτησε η κυρία Χολμάγερ. Δύο αφορούν την Επιτροπή Περιφερειών και μία την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Τις εξήτασα με ιδιαίτερη προσοχή και στις τρεις περιπτώσεις πρόκειται για το πλεόνασμα πιστώσεων από κάποιες γραμμές ιδίως για χαρτικά, ε, για υλικό γραφικό, γραφική ύλη μάλλον, και θα μεταφερθούν στην ε, ασφάλεια των έλεγχων των κτηρίων και την ασφάλεια των ε, τεχνολογικών μέσων έναν από τους στόχους που θέλαμε να ενθαρρύνουμε στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων έτσι κι αλλιώς. Προτείνω λοιπόν μετά από την εξέταση να τις εγκρίνουμε. Μας φαίνεται ότι η πίστοση και η μεταφορά της είναι λογική και εύλογη, εύλογο το αίτημα. Ε, βάσει του άρθρου 25 δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε εφόσον τα ποσά είναι ε, αρκετά χαμηλά οπότε αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θεωρώ ότι οι πιστώσεις αυτές, οι μεταφορές αυτές εγκρίνονται. Δεν υπάρχει κανείς που να θέλει να παρέμβει για την κτηριακή πολιτική. Στα διάφορα υπάρχει κάτι, δεν νομίζω. Οπότε σας επιβεβαιώνω ότι η επόμενη συνεδρίαση μας είναι στις 27 Οκτωβρίου 2017 και στις 12 Νοεμβρίου 2015 από 9 ως 12.30 και 3 έως 6.30 και στις 19 2015, ε, από τις 9 ως τις 12.30 ε, λήξη της συνεδρίασης Thank